για όλους σας. Σας ευχαριστώ κυρία Τζαβέλα και ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Το επόμενο θέμα έχουμε την αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σαρτόρη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το κείμενο αυτό προέρχεται από την Επιτροπή της οποίας προεδρεύω. Είναι συλλογικό έργο. Κατόπιν του ατυχήματος στη Φουκουσία πριν από δύο χρόνια. Στι ΔΕΑ 5 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφύσε την ανακοινωσή της όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων και την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τιμήσουμε τα θύματα όλων αυτών των πυρηνικών καταστροφών. Και γι' αυτό σήμερα στις ε, Δύο η ώρα στην Ιαπωνία τηρήθηκε ενό λεπτού σιγή και όλοι σταμάτησαν στις δουλειές τους. Το 2013, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Οδρή μπορείτε να εγκρίνει μια οδηγία όσον αφορά την πυρνική ασφάλεια και θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα και τούτης της συζήτηση, αλλά και τα ψηφίσματα που οποία μπορείτε να παρουσιαστούν και να υποβληθούν για ψήφισε την, ε, την ολομέλη αυτή, οπότε θα πρέπει να δούμε τώρα, υπάρχουν διάφορα σημεία, κάποια σημεία παιδιά και η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει βεβαίως να δούμε πώς θα βελτιωθεί η κουλτούρα, η αντίληψη για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει να μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιους κανόνες κοινού. Θα πρέπει να έχουμε διάδοση των καλύτερων ε, τεχνικών και εμπειριών. Και επίσης θα πρέπει να βάλουμε υπόψη τις ε, τεχνικές εκένωσης του χώρου μετά από ένα ατύχημα. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις ικανότητες του προσωπικού και επίσης να δούμε πώς θα έχουμε βελτίωση σε μια σειρά τομέων αλλά και στα όσα έχουν σχέση με την ασφάλεια και την ε, ανεξαρτησία των ε, αρχών που επιβλέπουν τις ενέργειας τον έλεγχο των δεδομένων που έχουν σχέση επίσης με τους πυρηνικούς σταθμούς. Θα πρέπει. Είπαμε. Οι συντονιστές της ε, Επιτροπής Ήτρε κατόπιν της ανακοίνωσης της 9 Οκτωβρίου είπαμε να πούμε ότι με αυτό μας το ψήφισμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη του Κοινοβουλίου. Προτείνουμε επομένω νομιμοθετικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν στον τομέα των πυρηνικών. Επ' αυτού τώρα θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα ζητήματα. Θέλουμε να μας βεβαιώσει ότι έχει λάβει υπόψη τα βασικά σημεία τα οποία αφορούν την ε, αναθεώρηση της νομοθεσίας για την πυρηνική ασφάλεια. Ε, για πες μας επίσης, θα προτείνει κάποια νομοθετικά κείμενα ε, τα οποία έχουν σχέση με την πυρηνική ασφάλεια πλευρά πολιτικών αρχών. Τώρα που έχουμε την υποβολή των προτάσεων. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι και οι εμπλεκόμενοι νομοθετικοί μηχανισμοί. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτά τα στοιχεία ασφάλειας μέσα στα πλαίσια της ενδεχόμενης χρηματοδότησης. Επίσης, η Επιτροπή θα αναλάβει κάποια δράση ε, για, ως προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και θα ισχύσουν οι συστάσεις ως προς τις διαδικασίες όπως ορίζονται στην ανακοίνωση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Σαρτόρη και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Πετινιέρ, στον Επιτροπό Πετινιέρ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τις, ε, τα τρομακτικά γεγονότα με το τσουνάμι που κόστισε όχι μόνο τόσες πολλές ανθρώπινες ε, ζωές και προκάλεσε τόσες ηλικές ζημιές, αλλά και προκάλεσε τόσο μεγάλες ζημιές στο πρινικό εργοστάσιο. Πολύ γρήγορα επιβάλαμε τα ευρωπαϊκά stress test. Ένα stress test που δεν είναι ένα stress test το οποίο εκ των προτέρων έπρεπε να εξυπηρετήσει το σκοπό του να επιβεβαιώσουμε δηλαδή ότι όλα πήγαιναν καλά στην Ευρώπη όμως το οποίο δεν θα ήταν και εκ των πραγμάτων αρνητικό αλλά το οποίο έπρεπε να είναι αντικειμενικό να καταγράψει το πώς έχει η κατάσταση από ασφάλειας των 135 πυρηνικών εργοστασίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ο σκοπό των stress test σε τρία επίπεδα. Για την χρήση των ε, εργοστασίων από τους εθνικούς ε, ε, φορείς από peer reviews σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου για πρώτη φορά ένας Αυστριακός συμμετείχε σε μια ομάδα στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή ένας Γάλλος στην Αυστρία, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών ε, εγκαταστάσεων. Η Ουκρανία, η Αρμενία και εκτός των Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή συμμετείχαν φορείς. Για κάποιου αυτό το stress test δεν ήταν αρκετά αυστηρό. Άλλοι το κρίνουν υπερβολικά αυστηρό στον Παρίσι, στη Βερολίνο, στην Πράγα δεν κάναμε καινούριου φίλους. Αντιθέτω. έχουμε πλέον τα αποτελέσματα στη διάθεσή μας και βάσει αυτών θα κάνουμε, τα λάβουμε τα περαιτέρω μέτρα μας. Καταρχάς, συμφωνήσαμε με τους εθνικούς φορείς να καταρτιστούν εθνικά σχέδια δράση για το τι θέλουν τα κράτη-μέλη, τι θέλουν οι ρυθμιστικές αρχές, τι θέλουν οι κυβερνήσεις βάσει των stress test που έγιναν στα κράτη-μέλη. Έχουμε πλέον τα στοιχεία μπροστά μας, αξιολογούνται και θα οδηγήσουν σε απαραίτητα μέτρα για τον ε, ε, νέο εξοπλισμό των ε, εργοστασίων. Κοιτάμε ποιες είναι οι νέες επενδύσεις που χρειάζονται και αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα πρινικά εργοστάσια. Αυτό θα κοστίσει 15 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά σίγουρα αυτό, το κόστος δικαιολογείται και έχει εξυπηρετεί ένα καλό σκοπό. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο α, μας κάλεσαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ανταποκρινόμαστε σε αυτό το κάλεσμα. Να ε, ξεκινήσουμε μια οδηγία για την πυρηνική ενέργεια στα τέλη Απριλίου θα παρουσιάσω στην, δημοσιότητα πώς θέλουμε να, να θεωρήσουμε την οδηγία για την πυρηνική ενέργεια, ποιες νέους όρους ε, θέλουμε να επιβάλλουμε, ποια είναι τα πορίσματα των ευρωπαϊκών stress test και τι θα σημαίνουν αυτά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτά θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αν γίνεται το επόμενο εξάμεινο. Προκειμένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της ε, στο Κοινοβούλιο, να λάβει την υποστήριξή σας και να ε, ζητήσει και την πλειοψηφία από πλευρά του Συμβουλίου. Ας μην αυταπατώμαστε. Η προθυμία στο Συμβούλιο για αποδοχή τέτοιων διατάξεων από την οδηγία πυρηνικής ενέργειας είναι πολύ διαφορετική. Πολλά κράτη-μέλη δεν θέλουν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να προδιαγράψει τα μέτρα ασφαλείας. Και θεωρούν ότι αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στην διαχειριτική ευχέρεια της κυβέρνησής τους, του Κοινοβουλίου της, του ρυθμιστικού της ε, οργάνου και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, στις μεταφορές, έχουμε προδιαγραφές ευρωπαϊκές που εξυπηρετούν τον πολίτη και θεωρώ ότι και σε αυτό το τομέα μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο ασφαλείας ευρωπαϊκό. Αυτό το χρειαζόμαστε. Μας ρωτήσατε, κύριε βουλευτέ, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας. Θα σας υποβάλουμε μια πρόταση μέσα στο έτος για δεσμευτικές ε, ε, διατάξεις για την προστασία των θυμάτων και ενδεχόμενων θυμάτων. Και προσανατολιζόμαστε σε πολύ διαφορετικές ε, ρυθμίσεις από αυτές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη σήμερα. Και σε ό,τι θεωρούμε ότι αξίζει από, από το εθνικό επίπεδο, θέλουμε να δώσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και επίσης έχουμε και διάφορα άλλες ε, ενδιαφέροντα ερωτήματα μπροστά μας. Ο συνάδελφος Αλμούνια για παράδειγμα. Θα διαπραγματευτούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού ενδεχομένω. κατά πόσον αυτό μπορεί να ε, δώσει εγγύησεις τιμών για νέα πρινικά εργοστάσια. Αυτό το θέμα δεν το ε, εξετάζω εθελοντικά. Αλλά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για μια νέα τέτοια market design. Αυτό θα είναι το νέο, η νέα λέξη το 2013 και η Βρετανική κυβέρνηση, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, θέλει να μας κάνει την εξή αίτηση. Θέλει και για τα εργοστάσια αερίου, αλλά και για τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, να έχει μία εγγύηση τιμής, προκειμένου Όποιο επενδύει σε νέα πυρηνικά εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα επόμενα 30 ε, έτη να έχει μια αγγιμένη ταρίφα, ένα αγγιμένη τιμή. Και η τιμή αυτή θα χρηματοδοτείται και από το Βρετανικό κράτος. Εγώ είμαι αρκετά διστακτικό σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση, αλλά περιμένω παρόμοιε προτάσει και από την Τσεχία και από τη Γαλλία, ίσω και από την Πολωνία. Επειδή όντω στέκει το εξή. Ίσως και από την Πολωνία, ναι. Γιατί όντω στέκει ότι στην παρούσα φάση σε πρινικά εργοστάσια στη Φιλανδία Κανείς δεν μπορεί να επενδύσει σε πυρηνικά εργοστάσια χωρίς κάποια εγγύηση τιμή. Το Μάιο θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο τέτοια ενεργειακά θέματα και κλείνοντα να πω ότι θεωρώ ότι το stress test μας ε, έφερε κάποια πορίσματα τα οποία δεν ήταν σίγουρα προηγουμένω σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις, τα θέματα ασφάλεια των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών και ελπίζουμε λοιπόν τα θέματα αυτά να τα συζητήσουμε στη δευτεροήμιση του τρέχοντο έτου με εσά και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Επιτροπέ Ούτενγκερ και τώρα κύριε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σήμερα και για να σας πω μετά τη συζήτηση για τις εκπομπές ε, αρίων θερμοκηπίου που θα κρατήσει μισή ώρα. Έχουμε 11 λεπτά. Θα πρέπει να ζητήσω λοιπόν από τους συναδέλφους ε, να δείξουν πειθαρχία. Η συνάδελφος Κουράσκα Μπομπίνσκα έχει το λόγο. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα τεστ αντοχής που ορίζει η νέα οδηγία αποτελούν ένα αγαστό παράδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια παρόλο που ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα κοινό αγαθό και άρα κοινό καλό. Σε σχέση με τα αποτελέσματα των stress test, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τους φόβους και τις αντιρρήσεις για τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρώπη είναι δραστήρια και ορίζει και δέχεται συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις όμορες χώρες. Μιλήσατε για την προσωμείωση στην Ουκρανία. Υπάρχουν όμως και άλλες χώρες που το προβλέπουν. Ίσως άλλες χώρες θέλουν να δημιουργήσουν λιγότερα δαπανηρές μεθόδους, γι' αυτό και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Κολάρος Καμπομίσκα. Και τώρα η συνάδελφος Μαντουρέλη για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πρώτα-πρώτα θα πρέπει να γνωρίσουμε... ότι αυτά τα stress test προϋποθέτουν ε, μία πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενο. Για άλλη μια φορά είναι πρωτοπόρα η Ευρώπη. Οπότε αυτή εξ αρχή αυτός ο εκούσιος χαρακτήρας α, και η έλλειψη της εξαρτησίας και αμεροληψίας για μας ήταν λόγος ανησυχίας. Και μόλις έγιναν ε, είδαμε ότι είχαν περάσει τις εξετάσεις ε, οι ποινικοί σταθμοί. Όμως ε, δεν έγιναν όλα σε Ευρώπη, γιατί επειδή εδώ πέρα τα θέματα επιδέχονται αμελητή κάποιες βελτιώσεις και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις, τι γίνεται με τις ε, απειλές που ακόμα δεν έχουν περάσει από αξιολόγηση Παρ' όλα αυτά, παρά τα θετικά αποτελέσματα να μην ξεχνούμε ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί κίνδυνο και γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ενέργειας ε, συγγνώμη, ε, ε, ασφάλεια το οποίο να μας εγγυάται την ασφάλεια. Και αυτό θα πρέπει να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι... Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ο συνάδελφος Τούρμη για μισή λεπτό. Ε, ε, Επίτροπε, αυτά τα stress test δυστυχώ είναι stress test τα οποία ε, επευλήθηκαν από την Γαλλία, από, την, ε, από το μεγάλο, τον Βασίλειο, εγώ στο από το Λουξεμβούργο να σας πω ότι αν συμβεί οτιδήποτε, μια ταμοκρατική ενέργεια κατά των εργοστασίων αυτών δεν θα πάψει να υπάρχει η χώρα μου. Ο δικός μου φόβος ποιος είναι, αυτά τα stress test να τύχουν κατάχρηση Και αυτό θα μας απασχολήσει στην Ευρώπη και γι' αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς είσαστε γνωστός για το εξή. Τους φορολογούμενους θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ειλικρινικά, με, ειλικρινά. Αυτό δεν ισχύει στην Ιαπωνία. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΠΚΟ, για παράδειγμα, ο φορολογούμενος τώρα πληρώνει το ατύχημα, το δυστύχισμα αυτό. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ασφάλειες. Ε, στις Βρυξέλλες θα αφήσετε ένα καλό όνομα ως επίτροπος αν φροντίσετε να υπάρχει να υπάρχουν ειλικρινές τιμές σε ό,τι, ειλικρινές ό,τι αφορά τις ασφάλειες. Δεν είναι δυνατόν να είναι πολύ μικρές αυτές οι ασφάλειες ή μη υφιστάμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε Τούρμες, το Σινόφσκι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι διότι τα τεστ αυτά κοπόσεως ε, λαμβάνουν υπόψη τόσο υψηλές προδιαγραφές και είναι ειδικά αυστηρού πλαισίου. Μετά από το ατύχημα της Φουκουσίμα θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι οι μονάδες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Ελπίζω η έκθεση αυτή να μπορέσει να άρει τις ανησυχίες που υπάρχουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να μην προσθέσουμε και νέα γραφειοκρατία. Επίσης βλέπουμε ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι πραγματικά αυτόνομες και υπήρξε αγαστή συνεργασία μεταξύ ΕΡΑ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πάσκα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 130 αντιδραστήρες που καλύπτουν το 34% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πυρηνικά έχουν εγκατασταθεί κυρίως στη Γαλλία, στη συνέχεια στη Σλοβακία και στο Βέλγιο. Γνωρίζουμε ότι το 1 τρίτον των ηλεκτρικών αναγών προέρχεται από πυρηνικά εργοστάσια και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθούν ατυχήματα. Επίσης, οι δοκιμές αυτές πέρσι δείχνουν ότι καμία, μας δική, καμία δική μας μονάδα δεν διατρέχει τέτοιους κινδύνους. Γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να μας πληροφορήσει τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να προωθήσουμε την ασφάλεια αυτού του ενεργειακού τομέα. Βίλς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μία δήλωση ε, πτώχευσης της ευρωπαϊκής πολιτικής μπροστά στους ευρωπαϊκούς ομίλου. Πριν από δύο χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως άλοθη ε, αυτό το σενάριο για τις stress test. Περίμενα ότι τουλάχιστον τα πιο επικίνδυνα εργοστάσια θα κλείναν. Αλλά φυσικά προτιμήσαμε το κέρδος επιπλέον. Βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση με την Ουκρανία για δύο πιστώσεις ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για την ε, συνέχιση λειτουργίας δύο Ουκρανικών αντιδραστήριων. Μετά την Φοκουσίμα και το Τσέρνομπιλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, ε, καλεί να αποκλείσουμε ένα νέο καταστροφικό σενάριο. Τα stress test θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για μια ευρωπαϊκή εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Ευχαριστώ, συνάδελφε Βίλτς. Ο συνάδελφος Βίλτσερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχεδόν σε όλα τα 135 εργοστάσια καταδείχθηκαν ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Και δεν έχουν λεφτεί καν υπόψη ενδεχόμενες τρομακρατικές ε, επιθέσεις. Μόνο Η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία μιλάει για αυτά τα 15 δισεκατομμύρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον ε, νέο εξοπλισμό των εργοστάσεων. Το σοκ της Φοκουσία μας λοιπόν καταδεικνύει ότι κανένα εργοστάσιο δεν είναι ασφαλές και όταν ε, η κάτοχοι και διαχειριστές των ε, πρινικών αυτών ε, εργοστασίων όχι μόνο δεν πληρώνουν, αλλά τελικά πληρώνονται για την ε, καθαρισμό μετά από τα πρινικά απόβλητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ελπίδη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, ο συνάδελφος Σίμπερ, όλοι ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν θα τα επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Επίτροπε, είπατε ότι δεν κάνετε φίλους το Παρίσι, στο Λονδίνο, με τα stress test. Μπορεί όχι στις κυβερνήσεις, αλλά μεταξύ του απλού κόσμου κάνατε φίλους. Εδώ πέρα ρόλος μας είναι να αγγιηθούμε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και νομίζω ότι ήταν σωστό βήμα λοιπόν τα stress test. Η πρινική ενέργεια είναι επικίνδυνη, είναι διασυνοριακή και γι' αυτό λογικά έπρεπε να είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν τα κράτη-μέλη. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Τούρμε. Μιλάμε για το επιχείρημα του κόστου. Αν κάνουμε μια πλήρη ανάλυση κόστου από αρχή μέχρι τέλου, καταδεικνύεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ ακριβή ενέργεια και θα πρέπει αυτή την αλήθεια να την προβάλλουμε. Γιατί είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προωθήσουμε άλλες ενεργειακές ε, μορφές, όχι αυτή την επικίνδυνη μορφή ενέργειας. Προφανώς ε, μπορούμε, πρέπει πάντα να, περιορίζουμε τις επιπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφος Φαμπρέμπτ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Δύο σημεία θα ήθελα να θίξω Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα stress test, είπατε κι εσείς ότι κάποιοι τα θεωρούν πολύ αυστηροί, κάποιοι λιγότερο αυστηρά. Το θέμα είναι τι απέφεραν αυτά τα τεστ. Στη δική μου χώρα κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι οι αντιδραστήρες ε, πέρασαν τα τεστ και μετά σε, έκθεση, σε μια έλεγχο ρουτίνας εντοπίστηκαν σφάλματα. διαπιστώθηκαν σχισμές ε, στους αντιδραστήρες. Αυτό κάτι λέει για τα stress test. Θα σας καλούσα λοιπόν να κάνετε ένα βήμα παραπέρα σε ό,τι αφορά την νομοθετική σας προσπάθεια. Για θέματα ευθύνη τώρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε μέχρι τέλους, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να τα ελέγχουμε όλα, διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε πλήρω την ενέργεια αυτή. Ευχαριστώ, συνάδελφε Φαμπρέμπτ, ο συνάδελφο Βλάσακ. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να θυμίσω κανέναν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος για όλα τα κράτη-μέλη. Και ε, νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μόνο τους αποφάσισαν να την διαθέσουν. Και έχουμε τώρα τις ρυθμιστικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε για την ασφάλεια. Σας συμμεθυμίζω επίσης ότι τα stress test για τους αντιδραστήρες ήταν ένα μέτρο το οποίο μετά την τραγωδία της Φουκουσίμα. Θελήσαμε να αξιολογήσουμε και πάλι την ετοιμότητά μας, την ε, στεγανότητα και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Τα stress test δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν την στάνταρ αξιολόγηση των αντιδραστήρων. Αυτή που γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Αυτό θέλουν τα stress test. Προ, προτείνονται επίση καινούριε ρυθμιστικέ αρχέ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό. Παρακαλώ, προσέξτε όμω, μην πολύ πολυνομοθετείτε, μην θεωρείτε ότι όλα κινδυνεύουν να γίνονται καλύτερα. Ξανααξιολογήστε τα πράγματα. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι όμορες χώρες ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες stress tests και δεύτερον σοβαρή διάσταση του θέματος που συζητάμε είναι η λειτουργία παραγωγικών σχολών εξειδικευμένου προσωπικού στις χώρες που λειτουργούν πυρηνικά εργοστάσια. στη φουκουσίμα είχαν τεράστιο πρόβλημα εξειδικευμένου προσωπικού όταν δημιουργήθηκε το δυστύχημα και δεν δεχόντουσαν αν θυμόσαστε καλά εξειδικευμένο προσωπικό να πάει από άλλες χώρες με το θέμα του περιβάλλοντος έχουν κλείσει όλες οι παραγωγικές σχολές που, μηχανικών ε, για τα πυρηνικά θέματα και πρέπει κύριε επίτροπε να το λάβετε σοβαρά υπόψη αυτό. υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον πυρηνικό τομέα. ευχαριστώ. Ο κύριος Ουρουτσέφ. Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ύπαρξης των ε, δοκιμών αυτό είναι επενεταίο και ιδιαίτερα επειδή οι μέθοδοι ήταν ενιαίες. Έτσι κατανοούμε καλύτερα τους κινδύνους που εμπλέκονται. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να βρίσκουμε λόγους αποκλειστικά επίκρισης. Οι δοκιμές ήταν ιδιαίτερα θετικές και υποστηρίζω το ψήφισμα που αναφέρεται στα μέτρα για να μπορέσουμε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως σε οτιδήποτε οδηγήσει σε υψηλότερες ε, τιμές ενέργειας. Αυτό είναι το λιγότερο που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να παγώσουμε τις τιμές αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Η ανακοίνωση της Επιτροπής ε, σε σχέση με την αξιολόγηση κινδύνων και ασφάλειας των ε, πυρηνοηλεκτρικών σταθμών δείχνει ότι θα πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις για την ασφάλεια των σταθμών αυτών. Επίσης, θα πρέπει να παροπλιστούν ορισμένοι σταθμοί και αυτό είναι μια δαπανηρή διαδικασία η αρχή του ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει το εμπλεκόμενο κράτος μέλος δεν είναι σωστή, ότι το εμπλεκόμενο κράτος μέλος είναι το μόνο υπεύθυνο, δεν είναι σωστή. Γιατί θα έπρεπε και οι όμορες χώρες να ασχολούνται, καθώς και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Γιόρταν. Κύριε Πρόεδρε, τα πυρηνικά είναι μεγάλος κλάδος. Είδαμε τι έγινε στην Ιαπωνία. Είδαμε πόσο σημαντική είναι το να υπάρχει επιτήρηση. Γι' αυτό και κάναμε τα στέστα. Δεν θέλουμε να απογορεύσουμε την πυρηνική ενέργεια. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε νέα μέτρα. Δεν εξασφαλίζεται έτσι η ασφάλεια. Αυτό πάντως που θέλω να ρωτήσω τον Ευρωβίτροπο είναι πώς βλέπετε τον ρόλο των διοικητικών αρχών σήμερα αλλά και στο μέλλον. Και τώρα διαδικασία Catch the και το λόγο έχει άλλο Τσάς. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι Επίτροπε, το... η έκθεση της καταστροφής της Φουκουσίμα πριν από δύο χρόνια σίγουρα μας άλλαξε σε ό,τι αφορά τις ε, ε, διαδικασίες ασφάλειας. Η απειλή της πυρηνικής ενέργειας δεν ε, επιτρέπει να μοιραστεί αυτή η ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών, γιατί μας αφορά όλους. Σε θέματα ασφάλειας και υγείας, η αρχή της πρόληψης είναι η πιο σημαντική. Αλλά τι γίνεται με τις αρχές μας όταν μιλάμε για αυτήν η ενέργεια. Η ευρωπαϊκή ενέργεια θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για μια απειλή για όλους μας. Χρειαζόμαστε συνεργασία πέρα από τα σύνορα και θα πρέπει αυτό να επηρεάσει όλες μας τις αποφάσεις θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τα προγράμματα ασφαλείας, αλλά να έχουμε διαμορφώσει όλοι μαζί αυτά τα προγράμματα ασφαλείας. Ελπίζω το ψήφισμα αυτό να μας βοηθήσει να κινηθούμε προς μια τέτοια κοινή ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε Κλάς, ο συνάδελφος Μπάνκι. Μικρό. Az Európai Unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági... ευχαριστώ πολύ. Σαν αφορά τους πυρηνικούς θερμοσυνέργειες, έχουμε κάνει τι δοκιμέ όπω έπρεπε και με επιτυχία. Και ο βασικό στόχο ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσον είναι αξιόπιστες συγκεντάσεις αυτέ ή ου. Ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλά επίπεδα στα οποία μπορούμε να ελέγξουμε την ασφαλειά του και ταυτόχρονα ότι όλα αυτά επιτελούνται από τα κράτη-μέλη. Στην Ουγγαρία, ξέρετε, Έχουμε κάποια ε, κεντρική αρχή στο ΠΟΤΣ και έχουμε ελέγχους οι οποίοι ασκούνται συνεχώς όσον αφορά την ε, ε, επιγραμμική προσβασιμότητα σε όλα τα δεδομένα. Έχουμε την Euratom, έχουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας που εμπλέκονται στο έργο αυτό. Και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εθνικές αρχές ε, επιτελούν αξιόλογο έργο και μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι οι ουγγρικές καταστάσεις ήταν από τις πιο ασφαλείς. Πάντως δεν χρειάζεται και άλλο ελεγκτικό επίπεδο παραπάνω. Ο συνάδελφος Ομπερμάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τα συστήματα ασφάλειας στη Φοκουσίμα ε, δεν ανταποκρίθηκαν λόγω του τσουνάμι, αλλά μετά την καταστροφή ε, έγιναν και τα stress test στην Ευρώπη. Σε 15 κράτη-μέλη τα τεστ αυτά καταδεικνύουν ότι χρειάζεται δισεκατομμύρια επένδυση για να ε, γίνουν πιο ασφαλή τα εργοστάσια. Το μοναδικό λογικό συμπέρασμα είναι ότι χρειάζεται να καταλήψουμε την πυρηνική ενέργεια σταδιακά και να προωθήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ακριβώ επειδή είναι ανυπολόγιστο το κόστο τέτοιων δυστυχημάτων. Πολλά κράτη ηγετικά, όπω η Γερμανία, αποφάσισαν να καταλήψουν την πυρηνική ενέργεια. Και το αντίθετο ερώτημα της ευθύνη σε περίπτωση ενός ατυχήματος και του μη υπολογιζόμενου κινδύνου. Και αυτό πραγματικά θα πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μάιερ. Και τώρα η συνάδελφος Μοκονάιτα. Ευχαριστώ, Επίτροπε, γιατί παρευρίσκεστε εδώ απόψε και σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία σας ως προς τις δοκιμές αντοχής στους πυρηνικούς σταθμούς. Ελπίζω η έκθεση να υπερψηφιστεί καταρχήν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πολύ υψηλά τον πύχη της ασφάλειας. Το κείμενο αντικατοπτρίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να είναι οι υψηλότερες δυνατές. Η Ρωσία και η Λευκορωσία θα πρέπει να διενεργούν τέτοιες δοκιμές γιατί διαφορετικά οι επιπτώσεις θα ήταν ολέθριες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαβουλεύσεις με τις γείτονες χώρες δεν προωθούνται. Σήμερα πανηγυρίζουμε την ε, εθνική μας επέτειο και ελπίζω να έχουμε υψηλότερες προδιαγραφές ε, ασφαλείας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την επέτειο την εθνική σας. Τελευταίος ομιλητή στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ευχαριστώ. Η καταστροφή της Φουκουσίμα ε, καταδεικνύει ότι πρέπει συνεχώς να ασχολούμεθα με την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, διότι διαφορετικά τα αποτελέσματα μπορεί να σταθούν ολέθρια. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αναλάβουμε μία συνεκτική προσέγγιση περί ελέγχων. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουμε άμεσα πυρηνικούς σταθμούς, αλλά χρειάζονται περαιτέρω, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση έτσι ώστε να έχουμε υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Η πυρηνική ενέργεια υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα 20% της ε, ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από εκεί, άρα θα ήταν κρίμα να κλείσουν οι στάθμοι αυτοί. Ο Επίτροπος Έτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να σας ευχαριστήσω για την πολύ αντικειμενική συζήτηση σήμερα το βράδυ και για τις συγκριτικές ε, που ε, ακούστηκαν για τα stress test και τα σχετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να σας πω ωστόσο ότι μεταξύ των εθνικών ε, φορέων και ημών τα stress test έγιναν βάσει εντατικής συνεργασίας με πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας ακόμα. Έχουμε ευρωπαϊκές ομάδες να ανταλλάξουν ε, εμπειρίες και τις τρέχουσες εβδομάδες οι επαφές είναι στενές για την πρότασή μας για μια νέα οδηγία για την πυρηνική ενέργεια. Μεταξύ άλλων, κοιτάζουμε και την αρμοδιότητα και την ανεξαρτησία των εθνικών υπηρεσιών. Κοιτάμε πώς ε, η επιτήρηση των, ε, σε εθνικό επίπεδο διαμορφώνεται και στο ιστορικό των Υπουργείων και εκτός των Υπουργείων. Κατά πόσον υπάρχει ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά δηλαδή την, ε, τους υπουργούς. Είναι διαφορετικά λοιπόν διαμορφωμένες οι αρχές εποπτείας στα κράτη-μέλη και θα ήθελα να πω ότι το υψηλότερο πρότυπο της ανεξαρτησίας ε, της υπηρεσίας εποπτείας θα πρέπει να αποτελεί τον ευρωπαϊκό κανόνα. Δεν χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία εποπτείας, αλλά θέλουμε κοινέ προδιαγραφέ ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώ θα γίνεται από πλευράς ποιότητα, από πλευράς ανεξαρτησίας αυτή η εποπτεία σε κάθε κράτο μέλος. Επιπλέον, η υποπτία στην Γαλλία είναι ιδιαίτερα υποδειγματική και ανεξάρτητη. και παρά την κριτική που αντιμετωπίζει, το stress test μας οδήγησε σε κάποια διαφωτιστικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία. Ξέρετε ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πιο πολύ πυρηνική ενέργεια από ό,τι ποτέ. Χρειαζόμαστε τέτοια διαφάνεια. Θέλουμε το άρθρο 194 να αποτελεί τη βάση για τις αρμοδιότητες. Η απόφαση για το πόσο θα χρησιμοποιείται η πρινική ενέργεια είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων και των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτό που εμείς ε, περιμένουμε, μάλλον τον Απρίλιο, δημοσιευτεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ασφάλειας και σε ό,τι αφορά θέματα ευθύνης και ε, αποζημίωσης θα σας υποβάλουμε μία πρόταση το Σεπτέμβριο. για ένα ελάχιστο καθήκον, ελάχιστο επίπεδο αποζημίωσης σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι σαφές ότι ο πλειοψηφία στο Συμβούλιο δεν θέλει να υπάρχει μια αυτόματη εγγύηση τέτοια. Στα εθνικά σχέδια δράσης ε, αποφασίζονται επενδύσεις ε, στα πρινικά εργοστάσια ύψους δισεκατομμυρίων. Και μόνο για αυτό το λόγο άξιζαν τον κόπο τα stress test, γιατί θα γίνουν τέτοιες επενδύσεις που θα εξυπηρετήσουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε αργότερα μέσα στο έτος για τις δύο οδηγίες και ελπίζω να υπάρχει υποστήριξη για μια μεγαλύτερη φιλοσοφία και νοοτροπία για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Επιτροπέ Oettinger. Και τέλος, ε, κατατέθηκε ένα ψήφισμα από την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας. Αύριο στις 12 θα ψηφίσουμε. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση και έχουμε μια κοινή συζήτηση για τις εκπομπές αερίων